So, welcome Καλώς ορίσατε όλοι στην κοινή συνεδρίαση των ε, Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων ε, και ε, Εσωτερικών Δικαιοσύνης και Ελευθεριών. Και είναι τιμή μου να συμπροεδρεύω με την Αντιπρόεδρο την κυρία Γκάλ. Ε, θα προεδρεύσει η ΕΚΟΝ στο, στην πρώτη έκθεση και η ΛΥΜΠΕ στη δεύτερη. Πρώτο θέμα, έγκριση μερίσιας διάταξης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 2 της ημερησίας διάταξης που είναι η εξέταση τροπολογιών της πρώτης έκθεσης πρόληψη της χρήσης του οικονομικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δύο εισηγητές έχουμε. Έναν από την Οικονομική Επιτροπή που είναι ο κύριος Κάριντς του ΕΛΚΑ και ε, ε, έναν εισηγητή που είναι εισηγήτρια από την Επιτροπή Ελευθεριών, η κυρία Σαρχεντίνη των Πρασίνων. Θα δώσω μέσα στο λόγο στον κύριο Καρίνς, τον οποίο και δεν βλέπω βέβαια. Ορίστε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, Chair. Uh, good morning to everyone. Happy New Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους όσους δεν συνάντησα μέχρι στιγμής. Ε, θα προσπαθήσω ε, για πολιτικός να μιλήσω σχετικά λίγο. Ε, για τις ε, τροπολογίες έχουμε περίπου 547 Ε, τα καλά νέα είναι ότι οι τροπολογίες δεν φέρουν επί του συνόλου του κειμένου αλλά επικεντρώνονται σε μια ομάδα ζητημάτων και ως εκ τούτου ε, είναι θεμητό να ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε καλή συμφωνία. Ε, ε, θα ε, εστιάσω την προσοχή μου σε τρία ζητήματα. Φαντάζομαι άλλοι θα θεωρήσουν ότι έχουμε περισσότερα ζητήματα. Θα τα σημειώσουν ούτως ή ούτω η άλλω. τελος παντων η καταχωρηση των ε, θα αρχίσω με τους δικαιούχους και την ε, καταχώρηση του σε μητρό. Πρόκειται για τις ε, τροπολογίες που αρχίζουν από 358 και μετά, άρθρο 28 και 30. Χρειαζόμαστε ένα νέο μητρό για τους δικαιούχους και νομίζω ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση περί αυτού. Βλέπουμε στις ε, τροπολογίες ότι υπάρχει μια μικρή διάσταση απόψεων ε, σε σχέση με το, ε, τη μορφή που πρέπει να λάβει αυτό το Μητρό. Έχουμε δύο οντότητες, τις επιχειρήσεις και τα καταπιστεύματα. Υπάρχει συμφωνία ότι χρειαζόμαστε δύο ειδών Μητρό. Προκύπτει και από τις τροπολογίες όμως ότι δεν είναι πλήρης η συμφωνία σε σχέση με το βαθμό προσπελασιμότητας ε, των ε, ε, μητρών, πρόσβασης μάλλον στα μητρώα. Τα μητρώα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν και για τις επιχειρήσεις και για τα καταπιστεύματα, όμως οντότητες όπως οι οικονομικοί ελεγκτές, οι κάτοχοι καζίνο, οι τράπεζες πρέπει να έχουν πρόσβαση, το ίδιο και οι αρμόδιες αρχές, φορολογικές αρχές, η κτλ. Θεωρούν όλοι ότι οι αρμόδιες αρμόδιες ε, αρχές ε, και όσοι υπάγονται στην υποχρέωση, τράπεζες και ούτω καθεξής, πρέπει να έχουν πρόσβαση. Τώρα, σε σχέση με τους περιορισμούς της πρόσβασης, υπάρχει μια μικρή διάσταση απόψεων. Κάποιοι θεωρούν ε, ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο οι επιχειρήσεις και οι μέτοχοί τους και άλλοι που θεωρούν ότι πρέπει να επιφυλάσσεται αυτό στα καταπιστεύματα. Είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε και στις συνεδριάσεις των σκιωδών. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη τις εγγνωμοδοτήσει των μεμονωμένων αρχών προστασίας των ε, προσωπικών δεδομένων. Ποιος είναι ο στόχος της οδηγίας. Είναι η καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από δραστηριότητες και η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ε, εφόσον μιλάμε για ε, δημόσια στοιχεία θα πρέπει να έχουμε περιορισμένη πρόσβαση ή δημόσια πρόσβαση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά τουλάχιστον δεν χρειάζεται χρειάζεται να συζητήσουμε αν χρειαζόμαστε μητρό, αν χρειάζονται ε, και για τι επιχειρήσει και για τα καταπιστεύματα, ε, είναι αν υπάρχει πρόσβαση μόνο για τι αρμόδιε αρχέ ή για του υπαγόμενου στην υποχρέωση. Αυτά έχουν κατοχυρωθεί ότι ε, χρειαζόμαστε ε, και τα δύο σε κάθε περίπτωση. Το θέμα μας είναι αν η πρόσβαση θα είναι μόνο για τι επιχειρήσει ή μόνο για τα καταπιστεύματα. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα, άρθρο 6, ε, τροπολογίες ε, που αρχίζουν από τη 245 και εφ' για την αποτίμηση του κινδύνου. Φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την αξιολόγηση κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν όμω κάποιε τροπολογίε και νομίζω θα πρέπει να τι συζητήσουμε ω προ το των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις εκτελεστικές ε, πράξεις ε, ως προς την ενίσχυση της νομοθεσίας όπου αυτό χρειάζεται. Ο κύριος Μπάλτσι, Γκίγκολτ και άλλοι έχουν καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Το εύρος των αρμοδιοτήτων λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις εφαρμοστικές πράξεις για την ευρωπαϊκό επίπεδο αποτίμηση κινδύνου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και δεύτερο ζήτημα, ε, ε, πώς, κατά πόσο θα δημοσιεύονται αυτές ε, οι αξιολογήσεις κινδύνου. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται και να γνωρίζει πού έγινε η μεγαλύτερη κίνδυνη. Όμως πόσο λεπτά θα το αλέσουμε, δηλαδή όταν μιλάμε για μια συγκεκριμένη χώρα, ορισμένες φορές ε, το κοινό είναι πιο ευαίσθητο σε σχέση με άλλα ε, ή σε άλλες ε, χώρες υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο επιχείρησης. Ένα καζίνο παραδείγματο χάρη. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες που είναι ευαίσθητες και εμπιστευτικέ, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα οπότε πρέπει να δούμε την κλίμακα δηλαδή εντάξει να δημοσιεύονται αλλά σε ποιο βαθμό να δημοσιεύονται σε ορισμένες χώρες ακόμη και στην Ευρώπη υπάρχουν κάποια τμήματα όπου υπάρχουν μεγαλύτερες μεγαλύτεροι κίνδυνοι κάποιοι παίκτε τη βιομηχανία, ακόμη και στο εσωτερικό ενό βιομηχανικού τομέα ή εμπορικού τομέα όπω τα καζίνο ε, ε, ελοχεύουν ιδιαίτερη κίνδυνοι οπότε θα πρέπει να δούμε το βαθμό πρόσβαση. Και τρίτον το πεδίο άρθρο 2, 10 τροπολογίε που αρχίζουν από την 178 μέχρι την 200 περίπου. Τώρα έχουμε τι τράπεζε του λογιστέ παρόχου ε, υπηρεσιών για τυχερά παιχνίδια και Όλοι πάγονται στο πεδίο ε, εφαρμογής της οδηγίας. Ε, κάποιοι ε, εισηγούνται την επέκταση του πεδίου, παραδείγματο χάρη οι εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, φυσικά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο, ε, είπανε κάποιοι, εγώ προσωπικά έχω κάποιους ενδιασμούς όταν μιλάμε για υπερευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η ΕΤΕ ε, αναρωτιέμαι ε, με ποιο τρόπο εμπλέκονται στην νομιμοποίηση σώδων από παράνομες δροσιτηριότητες ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες συγγνώμη αλλά θορυβούμε όταν το σκέφτομαι και μόνο τι σχέση έχουν ε, αυτά λοιπόν για τη διεύρυνση του πεδίου ή για την σμίκρινσή του, για τα τυχερά παιχνίδια παραδείγματος χάρη κάποια κράτη-μέλη ε, να ε, αποφασίζουν αν κάποιο είδους τυχερά παιχνίδια τίνουν προς την τέτοιου είδους νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες όχι μπορούν να αποκλειστούν από, τον, από την οδηγία, δηλαδή κάποια κράτη-μέλη μπορούν να πούνε ξέρω εγώ αυτό το μπίνγκο ας πούμε. Ε, εντάξει, εγώ δεν, στην πράξη δεν παίζω κιόλα. Ε, μία φορά το τόλμησα και έχασα 20 δολάρια και σταμάτησα να, να παίζω μετά. Ε, ε, κάποιοι ακούνε τη βιομηχανία τους, ε, τα στοιχήματα με τα στην Ιρλανδία παραδείγματο χάρη, πολλά λεφτά ε, και οι Ιρλανδοί περνάνε πολύ ωραία απογεύματα έτσι, εντάξει είναι σημαντικό για τις ντόπιες κοινότητες. Μπορεί η Ιρλανδική κυβέρνηση, λέω εγώ, να είναι σε καλύτερη θέση να αποφασίσει ε, στη θέση των Βρυξέλλων. Λοιπόν, ε, σμίκρινση μεγέθυνση του πεδίου, θα δούμε υπάρχουν επιχειρήματα ε, και από τις δύο πλευρές. Θα δούμε. Θα καταλήξουμε σε συνένεση φαντάζομαι για την προστασία των δεδομένων. Γίνονται σχόλια εκτός μικροφώνου, δεν τα ακούμε δυστυχώς. Α, ναι, μου λέτε ότι μιλάω γρήγορα. Να μιλάω γρηγορότερα ή πιο αργά. Τι λέτε εσείς. Ε, για την προστασία των δεδομένων δεν χρειάζεται να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, συνοψίζοντας θα έλεγα ε, ότι προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία με τους Κιώδης και δεύτερον ε, είναι καλές πιθανότητες που έχουμε να καταλήξουμε σε συνενετικές λύσεις και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε. Ε, μια συνενετική έκθεση του Κοινοβουλίου θα το φέρει στη δυνατή θέση για να εισέλθει διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ε, θα έλεγα επίσης ότι είναι καλό το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρώσουμε το έργο μας ε, και ή δυνατόν να ξεκινήσουμε και τις εργασίες μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ε, θητείας. Ευχαριστώ πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Κάρινσε. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Σατζεντίνη από του πράσινου που είναι η συγγήτρια Uh, Με βάση αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, θα ήθελα να σταθώ σε τρία ζητήματα. Καταρχήν ε, το μητρό αυτό για τους ε, δικαιούχους, τελικούς δικαιούχους και οι σοσιαλδημοκράτες, φλελεύθεροι και οι γκουέ έχουν υποβάλει αρκετές τροπολογίες καθώς και οι πράσινοι και το ΕΛΚ που ορίζουν ότι χρειάζονται αυτά τα δημόσια μητρώα και αυτό συμβαδίζει με τις προτάσεις των G8 και έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ε, να είμαστε πιο ανοιχτοί για το ε, τι κατέχουμε και τι οφείλουμε. Στην ιδιωτική μας ζωή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα προσβλέπω στις τροπολογίες συμβιβασμού που ορίζουν την ανάγκη δημόσιων μητρών. Αλλά αυτό είναι ανοιχτό ζήτημα που θα συζητηθεί με τον αποκοινού εισηγήτη. Το, το δεύτερο ζήτημα είναι η προστασία δεδομένων. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς σε σχέση με τις οντότητες αυτές και πρόκειται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καζίνο, ε, τράπεζες και ούτω καθεξής. Όλοι δηλαδή ε, που θα πρέπει να λογοδοτήσουν για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κύριος ε, Κάρενς και εγώ έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες για να συμβαδίσουν αυτά τα δύο νομοθετήματα και η Σοφή Ιντβέλτ έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες για την παρακράτηση δεδομένων. Νομίζω ότι χρειάζεται ε, κάποια διασάφηση και σε αυτό το τομέα. Η κυρία Μποσκουρτ και η κυρία Μακοβέη έχουν υποβάλει δύο τροπολογίες για την προστασία ε, όσων καταγγέλουν παράνομες δραστηριότητες. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι καταδότες και όχι καταδότες που να ορίζουν, να προωθούν πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες. Τώρα, το ερώτημα προς τους σκιώδεις είναι το εξής. Είσαστε ικανοποιημένοι με τη στάση των συνεισηγητών για την προστασία των δεδομένων γιατί έχουμε τροπολογίες από τη Σοφή Ιντβελτ και το Φρανκ Έγκελ από το ΕΛΚ που δεν συμβαδίζουν με αυτά που προτείνουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, το σκεφτήκατε, θεωρείτε ότι η πρόταση είναι επαρκής ή έχετε διαφορετική γνώμη. Τέλος. Ε, ο κατάλογος για τους ε, πολιτικά εκτεθειμένους, ο συνεισηγητής και εγώ θεωρήσαμε ότι πρέπει να αναθέσουμε στα κράτη-μέλη να ορίσουν αυτό τον κατάλογο όσων εκτίθενται ε, των δημόσιων προσώπων για τα δημόσια πρόσωπα. Και ο κύριος Βότσον ε, στην ουσία ε, μας είπε ότι εκεί που ε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να τα προωθήσουμε ιδιαίτερα για τα δημόσια πρόσωπα και τους συνεργάτες τους, για να ορίσουμε τα πρόσωπα αυτά σαφέστερα. Γι' αυτό ο συνεισηγητής και υποφαινόμενοι έχουμε τροποποιήσει την πρόταση Επιτροπής προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Τέλος, Έχουμε ε, μία συνάντηση σκιωδών την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο στις 6 η ώρα και για τις δύο επιτροπές. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αποσταλεί η ενημέρωση, αλλά να το λάβετε υπόψη για να δούμε που βρισκόμαστε και κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε συμβασμούς για να ακολουθήσουμε την όλη διαδικασία, να την επιταχύνουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρχεντίνη. Και τώρα πριν αρχίσουμε να ακούμε τους σκιώδες ηγητές. Ζήτησε το λόγο η κυρία... Όχι, δεν το ζήτησε. Ε, με τη σειρά τώρα σκιώδης από την Οικονομική Επιτροπή, πρώτος ο κύριος Σίμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, το θέμα των μητρών, αν θα πρέπει να είναι δημόσια ή όχι. Γνωρίζει η Επιτροπή ΕΚΟΝ ότι εμείς ε, θα πρέπει ε, να ζητούμε ε, να δικαιολογεί κάποιος γιατί ενδιαφέρεται, όπως ακτιματολόγια σε διάφορα υποθυκοφυλάκια κτλ. Ε, η μεγάλη πλειοψηφία όμως με έπεισε ότι είναι σημαντικό εδώ να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια ε, και να φαίνεται αυτό. Γι' αυτό είμαι υπέρ της δημόσιας ε, πρόσβασης για όλους, δηλαδή να είναι δημόσια τα μητρώα και να μην υπάρχουν περιορισμοί. Αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μόνο εκείνους που επωφελούνται από εταιρείες ανώνυμες, αλλά μπορεί να είναι τραστ, ε, καταπιστεύματα, ιδρύματα και άλλα ε, τέτοια μορφώματα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που ανέφερε ο εισηγητής της ΕΚΟΝ, εξαίρεση διαφόρων τομέων, ιδιαίτερα τα τυχερά παίγνια, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα ε, στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, ας πούμε το λότο στη Γερμανία, ε, με εθνική νομοθεσία ήδη από σήμερα ρυθμίζονται αυτά τα θέματα που σχεδόν αποκλείουν το ξέπλυμα χρήματος. Πάνω από 1000 ευρώ Οποιοδήποτε έμβασμα μπορεί να γίνει μόνο από τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό. Εδώ μιλούμε λοιπόν για ποσά κάτω των χιλίων ευρώ. Εξού και η πρόταση να υπάρχει αυτή η δυνατότητα μόνο αν τα κράτη-μέλη με συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι σε κάποιους τομείς δεν υπάρχει ε, κίνδυνος ή αμεληταίος, σε βάση περιπτώσει, για το ξέπλυμα του χρήματος. Και να ε, είναι πιο απλές οι ρυθμίσεις ή να εξαιρούνται. Ε, αυτό είναι θέμα του κράτους μέλους ε, το οποίο θα τα ρυθμίζει. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ή τα δημόσια πρόσωπα, ε, το είπα και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, έκανα μια πρόταση. Γνωρίζω ότι υπερβάλλει κατά πολύ το στόχο και αυτό που ζητάει η task force για τα χρηματοπιστωτικά, λέει είναι θέμα αρχής. Όταν μιλούμε για δημόσια πρόσωπα, για πολιτικούς, γιατί το αναφέρουμε αυτό. Διότι λέμε ότι εδώ υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πολύ σημαντικός ο κίνδυνος ξεπλήματος και είναι ιδιαίτερα τα προβλήματα ε, για τις χώρες, ε, για τα κράτη-μέλη, για την εσωτερική αγορά. Αλλά αρνούμε, αρνούμε και είναι προσωπική μου πεποίθηση ε, αυτό να το ε, ε, τονίσουμε και να το έχουμε αποκλειστικά και μόνο για πολιτικούς. Αν το γράψουμε αυτό δεν θα λέμε ε, στους Ευρωπαίους ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, αλλά να πούμε ότι τους πολιτικούς χρειάζεται να ελέγχουμε γιατί αυτοί χρειάζονται έλεγχο. Μα που γίνεται ξέπλυμα χρήματος στις τελευταίες δεκαετίες, ποιοι ενέχονται εκεί, στη δική μου χώρα ή και στην Ευρώπη γενικότερα. Για πείτε μου παρακαλώ, ας πούμε από τη Γερμανία να φύγω για να πάω στο Βατικανό. Και κοιτάξτε την τράπεζα του Βατικανού που τώρα την ε, ε, καθαρίζουν εκ βάθρων. Ε, τεράστια ξεπλήματα χρημάτων έχουν γίνει. Και γιατί οι εκκλησίες και οι διάφοροι ηθήνοντες εκεί και οι ιεράρχες να εξαιρούνται. Γιατί οι εξέχοντες επιχειρηματίες να εξαιρούνται. Συζητούμε μόνο για τους πολιτικούς, για δημόσια πρόταση. Ε, πρόσωπο. Τι συζητάμε τώρα. Πωλήσει όπλων. Γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα ε, που πληρώνουν μίζες ε, και τα εξετάζει τώρα η ελληνική δικαιοσύνη. Όλοι, όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν κάνει ξέπλυμα χρήματος. Και διερωτωμε με. Χώρες, ολόκληρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβλήματα με τη δράση ορισμένων εταιριών, οικονομικών παραγόντων. Κοιτάξτε τι κάνουν γερμανικές εταιρείες που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους στα έργα υποδομής, στα οικοδομικά έργα, ε, στις τρίτες χώρες, ε, οι κατασκευαστικές εταιρείες. Πολύ μεγάλες και ενδιαφέρουσες μεθόδους έχουν χρησιμοποιήσει για να πάρουν τα διάφορα έργα. Τώρα ε, όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι έχουν αλλάξει, αλλά έχουν ξεπλύνει χρήμα. Και διαρωτώ με γιατί να τους εξαιρέσω όλους αυτούς, για ποιο λόγο. Γιατί δεν διευρύνω τον κύκλο των δημοσίων προσώπων που χρειάζεται ιδιαίτερη ε, προσοχή. Μόνο η πολιτική είναι. Οικονομική ζωή υπάρχει δυσκολία, ε, ε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να λέμε ότι μόνο η πολιτική είναι. Δεν θέλω να εξαιρέσω κανένα, αλλά να βγούμε μόνοι μας και να πούμε ότι, α, κοιτάξτε, εμείς είμαστε αυτοί που χρειάζονται ιδιαίτερο έλεγχο. Δεν είμαστε. Γι' αυτό είμαι υπέρ πιο αυστηρών κανόνων και πιο σοβαρών ελέγχων και αυτό σημαίνει να μπουν και άλλα πρόσωπα που είναι δημόσια πρόσωπα και δεν είναι μόνο πολιτικοί. Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, αυτό που λέγεται PEPS με τα ε, αγγλικά αρχικά. Και ένα τελευταίο για την εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μία τριετία, μετά τη θέση σε ισχύ, θα πρέπει να εκπονήσει μία έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεταφέρει στην νομοθεσία του στα κράτη-μέλη τα μέτρα, τι κίνδυνοι υπάρχουν και τι μέτρα έχουν λάβει για να περιορίσουν τους κινδύνους αυτούς. Σημαντικό είναι αυτό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δηλώνουν τι έχει γίνει και να είναι υποχρεωμένα. Γιατί αυτό πρέπει να μπει στο κείμενο κατά την απόψή μας για να υπάρχει και ένας έλεγχος της όλης εφαρμογής και ε, της επιτυχούς εφαρμογής σε μια αναθεώρηση μετά από μια τρίτη όπου χρειάζεται αυτό και όπου είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέτερ. Και τώρα εξ ονόμα της Επιτροπής Ελευθεριών το λόγο έχει η κυρία Ποσκούρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. από την ομάδα μας και με βάση τις τροπολογίες βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα μητρώα δικαιώχων και τι μορφή θα έχουν. Νομίζω ότι οι πληροφορίες για τα μητρώα θα πρέπει, οι πληροφορίες θα πρέπει να υπάρχουν στα δημόσια μητρώα. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας αλλά θα πρέπει να δούμε ε, να είμαστε σίγουροι για το ποιες πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται Μιλάμε και για την προστασία δεδομένων των πολιτών. Αυτό το θέμα άπτεται της προστασίας των δεδομένων για τους πολίτες. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες για τα άρθρα 29 και 30 και ελπίζω οι εισηγητές να προβάλλουν τροπολογίες συμβασμού. Δεν θέλουμε να, να ψηφίσουμε παρόμοιες τροπολογίες γιατί θα αποδυναμώσουμε τη θέση μας. Εγώ έχω υποβάλει μία πρόταση για απαγόρευση εμπορικής χρήσης των καταλόγων που αφορούν τα δημόσια πρόσωπα, δηλαδή τις προσωπικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα και θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε. Επίσης να μπορέσουμε να ε, μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά για την νομιμοποίηση εσόδων και να έχουμε στοιχεία και για τους καταγγέλλοντες. Ως προς τα παιχνίδια τζόγου, κατανοώ αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν ε, μιλάμε για τυχερά παιχνίδια που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Γιατί αν το αφήσουμε στα κράτη-μέλη, τότε ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι τα στοιχήματα τύπου μπίνγκο ε, δεν ε, έχουν κινδύνους, ενώ ένα άλλο κράτος μέλος να έχει αντίθετη άποψη για τα ίδια τυχερά παιχνίδια. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση και επειδή το θέμα συζητείται μεταξύ κρατών μελών, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για στημένα παιχνίδια ή απάτες. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι καν ποινικό το, το θέμα αυτό, δηλαδή τα στημένα παιχνίδια και οι απάτες στον αθλητισμό, οι απάτες στον αθλητισμό. Αυτό δεν έχει ποινικοποιηθεί σε ορισμένα κράτη, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση. Θα φτάσουμε δηλαδή σε forum shopping και όσοι ασχολούνται με αυτή τη νομιμοποίηση εσόδων με βάση τα τυχερά παιχνίδια θα μεταβούν στα κράτη-μέλη όπου δεν είναι υπόλογοι και όπου δεν υπάρχουν κυρώσεις. Αυτά είναι τα σχολεία μου. Ευχαριστώ. Εξ της ΛΥΜΕ, ο κύριος Βάτσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την εξαιρετική τους εργασία. Χαιρόμαστε διότι πολλοί συνάδελφοι θέλουν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την προσέγγιση που βασίζεται στον πραγματικό κίνδυνο, ο οποίος βεβαίως διαφέρει και οποιοδήποτε κανονισμός θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος για να το λάβει αυτό υπόψη. Νομίζουμε ότι αυτή η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ε, δεν ε, ε, επιτρέπει δεν αφήνει πολλά περιθώρια στα κράτη-μέλη, απλώς θα πρέπει να γίνει καλύτερη στοχοθέτηση των οντοτήτων αυτών που νομιμοποιούν έσοδα παρανόμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη να γνωρίζουν τι κινδύνους διατρέχουν και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται αποτίμηση κινδύνου σε εθνικό επίπεδο και όχι ευρωπαϊκό. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή ε, ε, Αρχή ε, Τραπεζών θα μπορέσει να αντιμετωπίσει, θα μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι θα ήταν ευεργέτημα να ε, είναι διαθέσιμη ευρέως αυτή η αποτίμηση, αυτές οι αποτιμήσεις. Η προσέγγιση της Επιτροπής ε, δεν αφήνει περιθώρια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα τυχερά παιχνίδια και όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για νομιμοποίηση εσόδων. Δηλαδή υπάρχουν οντότητες ε, υψηλού κινδύνου και χαμηλού κινδύνου, γι' αυτό δεν μπορούμε να προβάλλουμε συνολικές λύσεις. Τα κράτη-μέλη θα ορίσουν ποιοι τομείς είναι υψηλό, υψηλού κινδύνου και ποιοι όχι. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει μία ε, συνολική, μία ενιαία προσέγγιση. Για να, πάρω για να δούμε ένα παράδειγμα. Ε, τα τυχερά παιχνίδια, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια. Ως προς τα παιχνίδια αυτά ε, online καταβάλλεται το αντίτιμο με πιστοτική κάρτα που έχει εκδοθεί από μία αρχή η οποία ε, έχει ελέγξει κατά πόσο υπάρχει τέτοια νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Δεν θα έπρεπε να γίνει το ίδιο, να γίνει μια ε, τέτοια αποτίμηση και από τον υπεύθυνο ε, τυχερών παιχνιδιών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας επιμερισμός στην αποτίμηση, γιατί μπορούμε να έχουμε αυτούς τους μικρούς γερανούς που τι κάνουν, ένα κουδάκι σε μία μηχανή όπου έχει βάλει, έχει σαγάγει κανείς ένα δίευρο ένα δίευρο, ένα νόμισμα. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση για αυτά τα μικρομηχανήματα με τα ε, καζίνο. Οι Φινλανδοί θέλουν να συμπεριληφθούν και τα slot machines, αλλά δεν ξέρω πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την χρήση και οπωσδήποτε χρειάζεται επικαιροποιημένη πληροφόρηση ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχουν κεντρικά μητρώα για τους δικαιούχους και τα οποία να δημοσιοποιούνται. Από πλευράς ήμανε ε, νομίζω ότι θα πρέπει να τύχει της ίδιας αντιμετώπισης σαν να πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο προϊόν, δηλαδή τα ε, το χρήμα που χρησιμοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της νομιμοποίησης. Ως προς τα personal equity plans θα πρέπει να ενταχθούν στον κανονισμό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία κατά του εγκλήματος μέσα στα πλαίσια της σταθερότητας και ολοκλήρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος και δεν θα πρέπει να έχουμε παρά ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει τις επιχειρήσεις να ανθίσουν μέσα όμως σε ορισμένα νόμια νόμιμα πλαίσια. Γι' αυτό έχουμε προωθήσει τις τροπολογίες 142 και 145 και θεωρώ ότι οι συγητές μέσα στα πλαίσια των τροπολογιών συμβασμού θα το δουν αυτό το ζήτημα. Θα συζητήσω με την κυρία Σαρτζεντίνη το θέμα της προστασίας δεδομένων. Και τώρα από την Επιτροπή Ελευθεριών θα δώσω το λόγο στον κύριο Κέρχοφ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Thank you very much, Chairman. I shall... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω κι εγώ κάποια πράγματα ε, για αυτό το ζήτημα, διότι είναι προφανές πως έχω αναλάβει το άλλο μισή της πρωτοβουλίας και σε λίγα λεπτά ε, πρέπει να μιλήσω για αυτό, οπότε θα είμαι και πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα, μην είστε πολύ καχύποπτοι σε σχέση με την ευελιξία που έχει ενσωματωθεί στην οδηγία. Τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν και αυστηρότερε διατάξει, χαμηλότερα όρια, το κρίνουν απαραίτητο. Πόσο ε, βασιζόμαστε στην αξιολόγηση κινδυνού, πρέπει να αλλάξουμε και την ονοτροπία όχι μόνο τη μέθοδο, και γι' αυτό ε, εισαγάγαμε αυτή την ευελιξία. Ε, η δημοσιονομική μονάδα δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλε αρμόδιε αρχέ Επίση είμαστε υπέρ τη προσθήκη, σε βάση της οποία τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ότι δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση και θα υποβάλλεται έκθεση για ύποπτε δραστηριότητε. Είναι πραγματικό ουσιαστικό ζήτημα η έλλειψη ανταλλαγή πληροφοριών, Κυρίω για του δικαιούχου. Θα πρέπει να δούμε ποιο τρόπο θα συνδεθούν πιο αποτελεσματικά τα εθνικά μήτρωα ή να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό ε, μήτρο. Εγώ μάλλον κλείνω προ τα εθνικά, αλλά τώρα με την κυρία Σαργιτζεντίνη, αυτό συζητάμε πολύ ε, εντατικά για τους ε, δικαιούχους. Ε, οι συγητές ελπίζουν να καταλήξουν σε μια εύκολα εφαρμόσιμη λύση. Τονίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα πρέπει ε, οι διεφθαρμένοι ή ε, οι εγκληματίες ε, να δυσκολεύονται λένε και περισσότερο να αποκρύψουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν. Για τα τυχερά παιχνίδια, όπως λέει και το Συμβούλιο, είναι ένας πολύ περίπλοκος τομέας. Να είμαστε λογικοί και ρεαλιστές όταν πραγματευόμαστε αυτό το ζήτημα. υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψε ανάμεσα στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου. Εγώ ήμουν και υπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήμουν ε, υπεύθυνο για αυτό το ζήτημα. Ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να επαφείται στην αρμοδιότητα του κράτου μέλου και η αποτίμηση γίνεται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, όπω σωστά είπε ο κύριο Βάτσον. Αφήστε που πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα στα ε, είδη των τυχερών παιχνιδιών, ε, υιοθετώντα την τελική μα προσέγγιση. Τέλο, θα χρειαζόμαστε με ρεαλιστικέ λύσει, βιώσιμε λύσει που θα λειτουργούν για του ιδιώτε που θέλουν να ανοίξουν ένα λογαριασμό, αλλά και για τι μικρέ, μεσαίε και μεγάλε επιχειρήσει ε, ε, θέλουμε να πιάσουμε τα μεγάλα ψάρια και όχι να δυσκολέψουμε τη ζωή των πολιτών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Κύρχοπ. Ε, από πλευράς της Γκουε δεν βλέπω κανέναν. Έχουμε ακούσει ε, τα μέλη των πολιτικών ομάδων, ε, μπορούμε ε, να περάσουμε στη γενικότερη συζήτηση. κυρία Γκυγιόμ, ζητώ συγγνώμη λέει η κυρία Γκυγιόμ για τη σύγχυση που προκάλεσα νωρίτερα επικροτούμε ε, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια ούτως ώστε να μειωθούν τα κίνητρα για την ε, οικονομική απάτη και το, την νομοποίηση εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Κατα, υποβάλαμε και εμείς τροπολογίες για πολλά και διάφορα ζητήματα που βλέπουμε ε, στο έγγραφο περιορισμός ε, των πληρωμών ε, σε ρευστό για τις ποινικές ακυρώσεις, για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου. Τέλος πάντων, να μην πολύ λόγο, τέσσερα στοιχεία θα ήθελα να σχολιάσω για τον περιορισμό των πληρωμών σε μετρητά. Θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπιστεί κάποια διάταξη για να αποφύγουμε την άγρα Δικαστηρίου το ε, Forum Shopping για ε, το ξέπλυμα χρήματος ε, για να μην επιτρέψουμε την εκμετάλλευση των πιο χαλαρών νομοθεσιών. Στη συνέχεια για τους ΠΕΠΣ, e τους πολιτικά εκτιθέμενους, θα έλεγα ότι τα, τα τρίτα κράτη και οι ΠΕΠΣ e έχουν ισότιμη μεταχείριση βάσει τη νόμου γάφη, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ω προ τη μεταχείριση που του επιφυλάσσουμε. Τρίτον, για την αποτίμηση κινδύνου τονίζουμε ότι η υπερεθνική μεταχείριση πρέπει με αποτελεσματικό τρόπο να εφαρμοστεί ε, από τα κράτη-μέλη, κυρίω όταν έχουμε στου ψηλότερου κινδύνου. Ε, για του ουσιαστικού δικαιούχου Τέταρτον, ε, βλέπουμε ότι οι εταιρείε σε βιτρίνα παίζουν κέριο ρόλο για το ξέπλυμα χρήματο, οπότε πρέπει να ξέρουμε ποιο ε, κατέχει, ποιος ελέγχει τις εταιρείες και ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ε, άρα χρειαζόμαστε ένα κεντροποιημένο μητρό προσβάσιμο στο κοινό με ε, τις απαιτούμενες και ουσιαστικές πληροφορίες για τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους. Αυτό είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος και αυτό ισχύει και για τα καταπιστεύματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει ένα ενίο μορφότυπο για ενιαία συλλογή δεδομένων Φερρυπίν και για την πρόσβαση των πληροφοριών εξάλλου ε, είναι προφανές ότι ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως ε, αυτά τα μητρώα συμμορφώνονται με τις ε, σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Ιδού εντάχει αυτά τα οποία ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστούμε κυρία Γκίγιον. Βίξτρομ και Σμιτ ακολουθούν. Thank ευχαριστώ. θέλω μόνο να εκφράσω την γνωμοσύνη μου προς τους δύο ε, συνεισηγητές ε, που εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα ε, να ασχοληθώ όλος ιδιαίτερος με την σημασία ύπαρξης των δημοσίων μητρών και από αυτό έχω καταθέσει και τροπολογίες για να μην επιτρέπουμε με την κατάσταση ε, ψευδεπίγραφων εταιριών ε, στην Ευρώπη είναι απαραίτητα. Ε, τώρα πρόσβαση για του δημοσιογράφους, για την κοινωνία των πολιτών, για το κοινό. Συνολική πρόσβαση χρειάζεται, ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να καταπολεμήσουν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες και να προστατεύσουν τους καταναλωτέ και να υποβοηθηθούν από τους καταναλωτέ για να εντοπίσουν στους όσους διαπράττουν αξιόπινες πράξεις, κυρίως σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, Αποφύγει μόνο προαγάγοντας ε, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ως προς ε, την ε, κατοχή των εταιριών. Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Οι ηγέτες της ομάδας G8 και οι ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφωνήσει ότι είναι κύρια σημασία να γνωρίζουμε τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και άρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις συστάσεις. Θα ήθελα παρακαλώ τους συνεισηγητές να λάβουν δεόντως υπόψη την σημασία σημασία ε, της, ε, των, δημοσίων ε, μητρών και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σμιτ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ευγνώμη προς τους συνεισηγητές και έχω ήδη μιλήσει για τη σημασία του κεντρικού και δημοσίου μητρώου. Θα ήθελα όμως να κάνω μια πιο προσωπική παρατήρηση. Ε, το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα ε, πρόβλημα που διαρκώς αμεγενθύνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με το, αυτά που συζητούμε εδώ. Ε, είδατε την περασμένη εβδομάδα ότι η βασιλική ισπανική οικογένεια εμπλέκεται σε τέτοιες δραστηριότητες, τουλάχιστον υπάρχουν βάσιμες υποψίες. Δηλαδή είναι ευρέως διαδεδομένο το φαινόμενο και δεν, λέω ότι δεν δεν πρέπει να παίζουμε τυχερά παιχνίδια, κάθε εβδομάδα παίζω εγώ αλλά υπάρχουν στημένοι αγώνες, υπάρχουν συνδικάτα ασιατικά μαφίας, ε, στημένα παιχνίδια σε μικρές ε, ε, κατηγορίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, πελώρια ποσά και χρησιμοποιείται εν μέρη αυτή ο διάβλος για ξέπλυμα χρήματος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει το πεδίο εφαρμογή να είναι διασυνοριακό. Μπορείτε να πείτε ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει τα στοιχήματα του υποδρόμου, όπως έλεγε ο προηγούμενος Επίτροπος μάλιστα. Ε, αρκεί αυτό. Ωραία. Και εγώ μπορώ να πάω στην Ιλάνδια να στοίχημα τη άλογα και ε, ε, μήπως ε, τίθεται ένα μικρό διασυνοριακό ζητηματάκι όπως και για τους ε, ποδοσφαιρικούς αγώνες. κάθε εβδομάδα συμβαίνουν αυτά. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε πιο αυστηροί και κάναμε αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή ΚΡΙΜ ή μήπως να την πούμε crime για, μιλώντας για το ξέπλυμα ε, χρήματος ε, παρακινώ λοιπόν ε, τους ε, εισηγητές να είναι λίγο πιο δραστηροί και να καταδείξουν ενισχυμένη θέληση, βούληση διεύρυνσης του πεδίου, κυρίως να αγγίξουν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και τον αθλητισμό, διότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας κάθε μέρα, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ τη δεκαετία του 60 δούλευα σε υπόδρομο, ήταν η πρώτη μου δουλειά. Έμαθα πολλά εκεί πέρα ε, πως ε, ήδη το 60 ξεπλέναμε χρήματα στον υπόδρομο. Προσοχή λοιπόν, ε, ελπίζω να ε, βάλετε τα δυνατά σας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούλινγκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή προέδρευσα την τελευταία φορά στη θέση σας ως πρεσβυτέρα στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, Θυμάμαι πολύ καλά τις συζητήσεις. Αλλά εμπιστεύομαι τον συνάδελφο Έγγελ ε, ε, που είναι σκιώδης ηγητής και Λουξεμβούργιο συνάδελφός μου για να τα πει σε λεπτομέρειες αλλά δυστυχώ σήμερα απουσιάζει. Εμπιστεύομαι πολύ και τον κύριο Κάρινς και πρέπει να πω ότι θα πρέπει πραγματικά να μην είμαστε εθεροβάμονες και σε αυτό το θέμα, να παραμείνουμε πολύ ρεαλιστές. Να σας πω δύο λόγια για το Μητρό. Είμαι υπέρ του Μητρώου και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα επιτρέψει στις τράπεζες ουσιαστικά που έχουν δυσκολίες ε, να βρουν τον πραγματικό ε, ιδιοκτήτη να κάνουν σωστά τη δουλειά τους στα πλαίσια ε, της καταπολέμησης ε, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είμαστε λοιπόν υπέρ του Μητρώου. Δεν φρονώ όμω ότι θα πρέπει να είναι δημόσιο αυτό το Μητρό, να έχουν οι πάντες πρόσβαση. Και οι δημοσιογράφοι, οι λομπί. Διότι πραγματικά ε, τότε μπορεί να προκληθούν προβλήματα και καταχρήσεις. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Ναι, λοιπόν, στην πρόσβαση όλων όσων ενδιαφέρονται και έχουν λόγο. Και είναι δημόσιες αρχές ή οποιοδήποτε άλλοι ε, έχοντες ε, κάποιο να αποχρώντα λόγο, αλλά όχι τελείως ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Επίσης, με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτό που ακούστηκε για τα δημόσια πρόσωπα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες δημόσια πρόσωπα, αμφιβόλου ηθικής αν θεωρούνται μόνο ε, αυτοί ως τέτοια πρόσωπο, θα έχει τεράστιες συνέπειες, σοβαρότατες αυτό. Γιατί αν υπερβάλλουμε εκεί, γιατί θέλουμε την πλήρη διαφάνεια και την απόλυτη, στα γερμανικά το αναφέρουν αυτός ο γυάλινος βουλευτής που είναι τελείως διαφανής κρίσταλο. Ε, τότε δεν θα βρείτε ε, άξιους ανθρώπους και ικανούς που να θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και να κατέλθουν στον πολιτικό στίβο. Δεν μπορεί να είναι όλα στο φως. Δυστυχώς έχουμε θλιβερά τέτοια παραδείγματα σε κάποιες χώρες. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με αυτό που είπε ο κύριος Σίμων προηγουμένως. Αλλά προβληματίζομαι και διαρωτώμαι ποια συνέπεια θα έχει αν γίνει δεκτή η τροπολογία 2.27 και 2.28 από τον εισηγητή του κυρίου Σίμων. Είναι και άλλες οι σημαντικές τροπολογίες, δεν θα τις αναφέρω για λόγους ωραχρονικούς, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Σε αυτά τα θέματα εμείς είμαστε σε ανταγωνισμό με τρίτες χώρες. Και θα ήθελα να μάθω τι ισχύει στις τρίτες χώρες για αυτά τα θέματα είναι φίλοι μας, εντάξει, φίλοι-φίλοι, αλλά και ανταγωνιστές. Και αν εδώ εμείς κάνουμε μια νομοθεσία η οποία αποθαρρύνει ακόμα και τους τιμίους και ειλικρινείς επενδυτές ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει προσοχή. Έχουμε μια τάση εδώ στο Κοινοβούλιο να επιβάλλουμε κανόνες, οι οποίοι πολύ συχνά τελικά διώχνουν τιμίους επενδυτές ε, ξένους γιατί υπερβάλλουμε. Λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω τι ισχύει παρακαλώ στις άλλες χώρες, τους ανταγωνιστές μας, για να κανονίσουμε την πορεία μας. Εσείς το βλέπετε αυτό ως πρόβλημα, το κατανοείτε. Μιλάμε και για θέσεις εργασίας, έτσι. Και τα καζίνο, δεν εργάζονται άνθρωποι εκεί. Εγώ δεν είμαι ειδική, ούτε εγώ είμαι ειδική. Μόλις χάσω 10 ευρώ στο Μοντόρφ Λεμπέν που έχουμε ένα ωραίο καζίνο εκεί στο Λουξεμβούργο. Α, πρέπει να σας πω ότι επί σειρά ετών ήταν ε, γορευμένο είδος αυτό, δεν υπήρχε καζίνο. Και τελικά άνοιξε γιατί υπήρχε ανταγωνισμός εκεί στη γύρω περιοχή. σε τρία, στα τρία χιλιόμετρα. Θυμάμαι ότι ήμουν εθνική βουλευτής όταν επιτέλους ε, δεήσαμε να κάνουμε μια παραχώρηση για ένα καζίνο στο Μοντόρφ. Λοιπόν, και μόλις χάσω 10 ευρώ εγώ σταματάω. Αυτό το θέμα λοιπόν του ανταγωνισμού το έχετε σκεφτεί. Ευχαριστώ πολύ ε, ε, και για τη συντομία σας. Θέλω να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα και σε αυτή όμως. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα εντάχει να ασχοληθώ με πέντε σημεία που εφήγησαν. Καταρχήν τα δημόσια ε, μητρώα ε, ιδιοκτητών ε, επιχειρήσεων και καταπιστευμάτων η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν μητρώα για αυτές τις οντότητες ε, δεν είχαμε όμως προτείνει μήτρο στην αρχική μας πρόταση, όμως ο Επίτροπος ε, κατέστησε σαφές ότι θα ήθελε να εισαχθεί ε, αυτή η έννοια των μητρών στην οδηγία και θα πρέπει να υπάρξουν και δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή ότι τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και επικαιροποιημένα και επίσης οι οντότητες αυτές θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως ποια είναι η κατάσταση του πελάτη τους. Σε σχέση με την προσβασιμότητα, Βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κάτι το οποίο θα καθοδηγήσει και τις συζητήσεις μας για τον βαθμό λεπτομέρειας των δεδομένων του Μητρώου. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο δεν εφήγει εδώ αλλά αφορά μία από τις τροπολογίες αφορά τον ορισμό των δικαιούχων, των απότερων δικαιούχων. Εμείς στην Επιτροπή, η Επιτροπή μάλλον, υπέβαλε μία πρόταση για τον ορισμό των δικαιούχων αυτών που συζητήθηκε στο Συμβούλιο και ε, δεχτήκαμε ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες ως προς τον ορισμό. Προβλέπεται ε, μία τροπολογία σύμβασμου από τον κύριο Κάριν. είναι 212, η οποία αντικατοπτρίζει την προσέγγιση του Συμβουλίου και θα την υποστηρίξουμε. Ένα τρίτο ζήτημα ε, σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια αναφέρθηκε, μάλλον η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε μία γενικότερη προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει όλα τα, τα τυχερά παιχνίδια, διότι οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο τα, τα καζίνο, όπως ε, όριζε η οδηγία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Συμφωνούμε λοιπόν με τα σχόλια που προαναφέρετε, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες αναλογικά και προβλέπουμε και τη δυνατότητα ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να παρεκκλίνουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως αν υπάρχει χαμηλός κίνδυνος. Ως προς την αποτίμηση κινδύνων, ε, αφορά ένα βασικό στοιχείο της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο η Επιτροπή θα μπορούσε να δεχτεί μια συντονισμένη προσέγγιση, όμως ε, δεν μπορεί να τα καταφέρει από μόνη της. Θα πρέπει οι εμπειρογνώμονες των ε, κρατών μελών, καθώς και της Επιτροπής, να συνδράμουν με βάση το input της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας και με βάση τις εθνικές αποτιμήσεις κινδύνου. Για την προστασία δεδομένων η Επιτροπή δέχεται την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη στεναρή θέση. Αυτή όμως θα πρέπει να προβάλλουμε μία ισόρροπη προσέγγιση έτσι ώστε να μην αντιταχθούμε στην οδηγία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Για λόγους συνέπειας θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε ε, τα κείμενα για την προστασία δεδομένων και να μην ε, πολλαπλασιάσουμε αυτά τα ε, κείμενα, τα οποία δεν βοηθούν για θέματα νομικής ασφάλειας. Για την περίοδο κράτησης των δεδομένων παρακράτησης των δεδομένων, δεν θεωρούμε ότι η διετής αυτή η περίοδος είναι επαρκής και οι οργανισμοί πληροφόρησης δεν θα μπορούσαν να μας δώσουν το κατάλληλο feedback. Και άρα τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν πρόωρα να καταστραφούν. Θα πρέπει να δούμε το όλο θέμα κατά περίπτωση για την παρακράτηση των δεδομένων πέρα από αυτή την προθεσμία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τέλος θα δώσω το λόγο σε, στους δύο εισηγητές, Κάρινς και μετά Σαρτζεντίνη. Θα ήθελα να είσαστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι θα λύσουμε το θέμα ε, με βάση την κατάχρηση στον τομέα της φοροδιαφυγής αν έχουμε μόνο αυτή τη μονομερή προσέγγιση. Στόχος είναι ο, αυτός που εγκληματεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες και ο νομιμόφρον από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση. Δηλαδή θέλουμε να πατάξουμε τους εγκληματίες και όχι να ε, καταστήσουμε τη ζωή δυσκολότερη για τους ε, νομοταγείς. Διότι το 95-99% των επιχειρήσεων δρά ε, νόμιμα ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των ΜΜΕ. Έχουμε πολλές ΜΜΕ που απασχολούν 10 άτομα και μόνο. Αυτό αφορά τη δική μου χώρα που έχει σωρία τέτοιων επιχειρήσεων, το 90-95%. Ε, αυτές οι επιχειρήσεις δεν ξεπλένουν βρωμικό χρήμα, είναι σαφές αυτό. Άρα έχουμε μια πολύ καλή βάση για συζήτηση. Αυτά που είπε ο Πέτερ Σιμών για τις τροπολογίες του 2.25 μέχρι 2.28. Ο, αυτός που εκτίθεται πολιτικά, ο πολιτικός δηλαδή, ε, βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ομάδας υψηλού κινδύνου για καταχρήσεις και διαφθορά γιατί ο πολιτικός μπορεί να υποβοηθήσει μία ε, επιχείρηση, επιχειρήσεις, ε, διαδικασίες εκχωρήσεων και ούτω καθεξής. Όμως, λάβετε υπόψη μία μεγάλη πολυεθνική, την IBM, τη, τη Siemens, ο, ο διευθύνων σύμβουλος αυτών των επιχειρήσεων έχει λιγότερη ε, ισχύ από μια ομάδα πολιτικών γιατί ξέρουν τι θα πουλήσουν, πώς, γιατί, ε, πώς θα διακινήσουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν το πεδίο δράσης ε, για άλλους. Δηλαδή θεωρητικά υπόκεινται είναι εκτεθειμένοι σε διαδικασίες διαφθοράς, αλλά η πολιτική είναι πιο ευάλωτοι γιατί μπορούν να δράσουν στο πεδίο δράση, εκεί δηλαδή όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή εμείς είμαστε πιο εκτεθειμένοι. Μιλάμε για ε, αυτούς που κατέχουν πολιτική, διοικητική ή επιχειρηματική θέση. Δεν νομίζω ότι η ιδέα στη βάση της είναι λαθανσμένη, αλλά αν ανοίξουμε αυτά τα παραθυράκια, τότε ε, θα μπορέσουμε να δράσουμε υπερβολικά και να πλήξουμε και τους νομιμόφρονες. Οι τροπολογίες σας είναι πραγματικά καινοτόμες. Στην αρχή είπα, είναι παράλογες, μετά είπα ναι είναι λογικές, αλλά πώς μπορούμε να, να τα διατυπώσουμε ακόμα καλύτερα. Θα σταματήσω όπως μου είπε ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Κάρινς, η κυρία Σαρτζεντίνη. Ε, πάντα ακούω πολύ προσεκτικά δύο θέματα. Καταρχήν το δημόσιο μητρό. Ας είμαστε σαφείς, απόλυτα σαφείς. Όταν μιλάμε για δημόσια μητρώα ή δημόσια πρόσβαση στα μητρώα αυτά των πραγματικών δικαιούχων, θα θέλαμε να ξέρουμε ότι τα μητρώα εμπεριέχουν τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες. Γιατί θέλετε να προστατεύσετε τους ανθρώπους που εντάσσονται σε αυτά τα μητρώα αλλά και γενικότερα από πλευράς αρχής ε, προστασίας δεδομένων δεν συλλέγεται στοιχεία που δεν χρειαζόσαστε για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή είναι μια γενική αρχή και με βάση αυτή την αρχή μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς ως προς το Μητρό. Χαίρομαι επίσης διότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ τάχθηκε υπέρ των δημοσίων μητρών, ε, τα οποία θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτό είναι ένα ε, ζήτημα τεχνικής υφής που θα πρέπει να επιληθεί μόλις ε, ληφθεί η απόφαση εισαγωγής αυτών των μητρών. Δεν μπορούμε να πούμε ας το ξεχάσουμε διότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να κρατήσουν αυτά τα μητρώα επικαιροποιημένα. Συμφωνώ με το άλλο αίτημα. Εάν υπάρχει δημόσιο μητρό, δεν σημαίνει ότι η έρευνα αυτή από τις υπόχρες οντότητες δεν θα γίνει. Οι υπόχρες οντότητες θα πρέπει να ε, γνωρίζουν ότι τα στοιχεία που διαθέτουν είναι τα σωστά. Τέλος, αυτή η οδηγία ε, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ε, δραστηριότητες είναι μία πιο ε, σωστή αντιμετώπιση για να πιάσουμε τους εγκληματίες, αλλά δρούμε σε εθνικό επίπεδο, γι' αυτό και το θέμα των τυχερών παιχνιδιών δεν έχει αντιμετωπιστεί. Νομίζω λοιπόν ότι διαφέρει από χώρα σε χώρα, εκεί δηλαδή που υπάρχει ο κίνδυνος στα τυχερά παιχνίδια επιγραμμικά ή Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σαρτζεντίνη και ζητώ συγγνώμη. Θα ψηφιστούν θα ψηφιστεί η έκθεση στις 22 Ιανουαρίου από την ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ. Και δίνω το λόγο στην κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσουμε με τον κανονισμό για την ενημέρωση για την μεταφορά ε, πιστώσεων. Ο Πίτερ Σίμεν και ο κύριος Κύρχοπ είναι συνεισηγητές. Ε, έχουμε μόνο 20 λεπτά στη διάθεσή μας, συνάδελφοι. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Οι συνεισηγητές θα έχουν 5 λεπτά έκαστος. Θα είμαι πολύ αυστηρή. Μετά θα έχουμε τρεις κοιόδης, Μήτρας, Μποσκούρτο και Σαρτζεντίνη. Εκείνοι θα μιλήσουν 2 λεπτά έκαστος και ε, οι συνάδελφοι που θα θελήσουν στη συνέχεια να παρεύουν μετά τους ε, σκιώδεις, ε, ρωτάω τώρα, υπάρχει κάποιος. Εάν όχι, κλείνω τον κατάλογο, κανείς δεν θα μιλήσει μετά. Θα ακούσουμε μόνο τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζήμων. Sorry, sorry, Mr. Peter Simon. Sorry, sorry. Ja, herzlichen äh, äh, ähm, Uh, Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη από την ε, Μόια ε, που δεν μπορούσα να... ζητά συγγνώμη η Μόια που δεν μπορούσε να έρθει αλλά γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Μόια. Θα την ενημερώσω για τα πεπραγμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ε, υπέβαλαν τροπολογίες, ε, καθώς και τον συνεισηγητή, τον κύριο Κύρκο, ε, διότι εργαστήκαμε με αγαστό τρόπο. Ε, συνεργαστήκαμε μάλλον με αγαστό τρόπο. Οι περισσότερες τροπολογίες ακολουθούν την κατεύθυνση που ακολουθεί και το σχέδιο που εξετάζουμε και επικροτώ την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων μέσω των τροπολογιών που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι. Βεβαίω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των εμβασμάτων ε, στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε διαφοροποιήσεις ε, ε, για τους ελέγχους εμβασμάτων που συνδέονται ή δεν συνδέονται με λογαριασμούς και γενικότερα μεταφορές πιστώσεων που συνδέονται ή δεν συνδέονται με τραπεζικούς λογαριασμούς στην ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να μην ε, δημιουργηθούν νέε αιστείες εγκληματικής δραστηριότητας και γι' αυτό ε, σε περίπτωση ανεξαρτήτων εμβασμάτων που δεν συνδέονται με τραπεζικό λογαριασμό θα υποχρεούται ο κάτοχος ε, του συστήματος να εξακριβώσει τα στοιχεία και, του, ε, ε, και αυτού που πραγματοποιεί το έμβασμα και του αποδέκτη, του απολύπτη και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν επαρκή στοιχεία και για τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση ε, για τις μεταφορές που γίνονται εντός και εκτός αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνεί με τον ε, ε, εισηγητή σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων για τις μεταφορές στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι επαρκούν αυτές τις πληροφορίες πιστεύει και ε, ε, επιτρέπουν την εξακρίβωση και τον εντοπισμό. Δεν χρειάζεται να θεσπίσουμε άλλες υποχρεώσεις διότι αυτό αντι Στου ε, στους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτά είπε η Μόγια και πάλι συγχαρητήρια. Ε, ελπίζω να επανέλθει εγκαίρως ώστε να ολοκληρώσει ε, αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε και από εμά συγχαρητήρια προς τη Μόγια. Ο κύριος Κύρκοπ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, αρχικά να ευχαριστήσω την συνεισηγήτριά μου και να την συγχαρώ για το ευχάριστο γεγονός. Ε, νομίζω ότι με σημειώθηκε αρκετή πρόοδος ε, και ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει σημειωθεί ακόμη μεγαλύτερη. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιο ε, είναι το ζήτημά μας, ποιο είναι το βασικό θέμα. Ε, θέλουμε να εντοπίζουμε ε, πιστώσεις και άρα επιβάλλουμε υποχρεώσεις για τις πληροφορίες, τις συνοδευτικές πληροφορίες για να μπορούν να διεξάγονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Μέσα σε αυτό το πακέτο βάσει του τωρινού καθεστώτος παρατηρείται μια μετατόπιση προς προσέγγιση που βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου και είμαι υπέρ αυτού. το, τα πρότυπα FATF λειτουργούν ως σε γραμμές ε, σε αυτό το τομέα και δεν χρειάζεται εμεί να επανεφεύγουμε τον τροχό. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιτυχή, ε, διότι ουσιαστικά μεταγράφει του κανόνε ε, τη ΦΑΤΦ. Όμω ε, υπάρχουν και κάποια ζητήματα συμφερόντων κρατών μελών. Ε, Εντάχει να τα ε, θίξω. Πρώτα απ' όλα το όριο. το όριο των χιλίων ευρώ που είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παραμείνει ακέραιο. φυσικά η ευελιξία έχει ενσωματωθεί ούτω ώστε οι μεταφορέ πιστώσεων κάτω του ορίου που παρόλα αυτά δημιουργούν υποψίε μπορούν να υπαχθούν σε οικονομικό έλεγχο. Ε, τροπολογίε τροπολογίες για τον κανονισμό ε, κονδυλίων αναφέρουν αυτή την υποχρέωση όταν ε, συμβαίνουν οι μεταφορές στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΦΑΤΦ ε, ζητά την, ε, δέχεται συγγνώμη, την τωρινή προσέγγιση, διότι ακολουθεί το γενικευμένο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του ξεπλήματος χρήματος. το άλλο ζήτημα είναι η άμβλυνση του ανταγωνισμού ως προς τα αισθήματα μεταφορός, μειώνοντας το άχθος για τους φορείς, μειώνοντας το διοικητικό άχθος και ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να προσφέρουν ε, να κάνουν πιο ανταγωνιστικές προσφορές ε, κυρίως ε, για χαμηλότερα ποσά. Οι καταναλωτές επίσης δεν θα χρειάζεται να επιβαρύνονται τόσο πολύ για να κάνουν μεταφορές μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91 και 92 τροπολογίες κτλ. που έχει καταθέσει ο κ. Γκοζές και η κυρία Γκουλάρα μας βρίσκουν σύμφωνα. σε 51, 52, 53 που έχει καταθέσει Ιντεβελντε και Σατζεντίνη, Ταβάρε και ο κύριος Τριανταφυλλίδη ε, απαλήθουν ε, την αναφορά στην αιτιολογική σκέψη παριθμών 7 στην οδηγία 4556 ε, ΕΚ για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την ευαισθησία των πληροφοριών. Επιτρέπονται έτσι μεταφορές προς τρίτες χώρες, όμως εκεί δεν κατοχυρώνεται επαρκέ επίπεδο προστασία των κοινών συμφερόντων ε, ή για την παροχή πληροφοριών για τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεων. Έχω καταθέσει και εγώ τροπολογίες ε, σε σχέση με αυτή την, ε, αυτό τον κανονισμό προστασίας των δεδομένων, διότι αυτό επηρεάζει τις σχέσεις παρόχου με καταναλωτή και η συλλογή προσωπικών δεδομένων για το ξέπλυμα χρήματος λαμβάνει η χώρα ταυτόχρονα με την συλλογή στοιχείων για εμπορικούς σκοπούς. Για να γίνονται σεβαστά τα ατομικά δικαιώματα είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι οι υποκείμενοι του δικαίου ενημερώνονται δεόντω ε, και άρα ε, κατοχυρώνονται τα δικαιώματά του ω προ την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν νομίζω να θέλω να πω τίποτα άλλο. Ε, θα σταματήσω εδώ. Ε, προσβλέπω στη μελλοντική μα συνεργασία για τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε. Είμαι αισιόδοξο. πιστεύω θα τα καταφέρουμε και στο μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη τις απόψεις και τα αιτήματα των υπολείπων. Ευχαριστώ. Περνούμε στους σκιώδεις Έκον Έλκ Νίτρας. Παρακαλώ. E, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα πω όλα σε δύο λεπτά, να συνοψίσω. Στις δικές μου τροπολογίες έχω εστιάσει κυρίως στα βασικά στοιχεία. Κυρίως πρόκειται για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και ε, για τις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα να σας εψίσω προσοχή στην τροπολογία υπαρθμών 72 που θέλω να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού έτσι ώστε να ε, καλύπτει ε, και ε, άλλα πεδία της αγοράς. Το άρθρο 3 δεν καλύπτει τα νομικά πρόσωπα από την άλλη. Ε, ε, Με μεγάλο ενδιαφέρον ε, διάβασα ορισμένες τροπολογίες και πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες βαίνουν στην ίδια κατεύθυνση, πράγμα που είναι υπέρ της ενισχυμένης προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ενημέρωσής τους. Είναι σημαντικό αυτό ε, στην ε, διαδικασία επεξεργασίας ή στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων και επίσης εδώ έχει σημασία ο νέος αριθμός ε, αναγνώρισης ή ταυτοποίησης. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένες επιμέρους λύσεις, αυτά που έχουμε στην τροπολογία Γκίκολ Ταβάρης και Αργεντίνης στην 125 δηλαδή, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή μεταξύ κρατών μελών να υπάρχει κάποια αντιστοιχεία των νομικών συστημάτων. Δεν είμαι βέβαιος ε, καθόλου ε, πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό και να εξασφαλιστεί, μας περιπτώσει. Και πώς μπορεί να επεκταθεί μάλιστα και σε χώρες που δεν έχουν αντίστοιχα με τα δικά μας συστήματα ή ανάλογα. Χαίρομαι που ορισμένα μέλη είναι υπέρ της απλουστευμένης πληροφορίας. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει πάντα το όνομα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν το άρθρο 5 δεν υπερβάλλει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης ε, από τη Λίμπε και τη σοσιαλιστές η κυρία Μποσκούρτ. Με ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε την προσέγγιση της συγκήτριας κυρίας Κλέβα, όπως είπε ο κύριος Σίμων. Ε, ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ. Η κυρία Σαρχεντίνη, σκιώδης των Πρασίνων από την Επιτροπή Ελευθεριών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κίρκοπ, τον δικό μας εισηγητή και της κυρίας, ε, την κυρία Κλέβα που ήταν εισηγήτρια από την ε, Οικονομική Επιτροπή. Θα πρέπει ε, επίσης να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου Ρουί Ταβάρης, που είναι ο σκιώδης του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, από τα εξή δύο, να τονίσω ιδιαίτερα. Εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ε, η δυνατότητα να ταυτοποιείται πλήρως και ο καταβάλλον ε, το ποσό αλλά και ο αποδέκτης όπως αναφέρει στην ε, τροπολογία 70 να ξέρουμε ποιος είναι και ποιος είναι ο τραπεζικός λογαριασμός του και αυτό έχει να κάνει και με την καταπολέμηση τροποκρατίας και την καταπολέμηση νομοποίησης εισόδων από παρανόμες δραστηριότητες. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Να το πω αλλιώς διαφορετικά πρώτα. Ο κύριος Κέρκοπ έκανε κάποια σχόλια για την τροπολογία 51, όπου διαγράφουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε ε, δεδομένα στο εξωτερικό σε τρίτες χώρες, οι οποίες δεν έχουν τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας αυτό το θέμα είναι κρίσιμο, διότι θα υπονομεύαμε όλες τις προτάσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων αν επιτρέπαμε να αποστέλλονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής ένωση σε χώρες που δεν συμμορφώνονται ε, με τους δικούς μας κανόνες για την προστασία. Γι' αυτό έχουμε κάνει και την τροπολογία 52 σχετικά και βλέπω ότι η συνάδελφος Σοφή Νετσφέλτ έχει κάνει ακριβώς το ίδιο στην 51 τη δική της. Για να πετύχει λοιπόν αυτή η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, επαναλαμβάνω, να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα και για την προστασία δεδομένων αλλά και για τους καταγγέλλοντες ε, και θα κάνουμε περαιτέρω τροπολογίες από αυτό. Ευχαριστώ κυρία Σαρχεντίνη. Δεν είναι παρόντες άλλοι σκιώδης ηγητές, ούτε άλλος βουλευτής έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα σύντομος και να απαντήσω στα σημεία που εφήγησαν. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια με την οδηγία για τις υπηρεσίες καταβολής πληρωμών. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ως προς την ορολογία και ιδιαίτερα προσεκτικής, γιατί στην οδηγία ε, περιπληρωμών δεν ενέχονται όλα τα στοιχεία που θέλουμε να εισαγάγουμε στον κανονισμό. Ιδιαίτερα την αντικατάσταση του ενιαίου, ε, ενιαίου, της ενιαίας οντότητας συναλλαγών του αριθμού σήμανσης της συναλλαγής με ένα ενιαίο σύστημα αντιμετώπισης των συναλλογών. Και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ορισμένες δυσκολίες ως προς τη συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές ως προς τις επαληθεύσεις των συναλλαγών κάτω των χιλίων ευρώ, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι αυτό σημαίνει ότι η διαβίβαση των δεδομένων θα διονγκωθεί και με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα δεν θα πρέπει ίσως να γίνει αυτή η διόγκωση. Εκφράστηκε η ανησυχία ότι χωρίς αυτό το κατόφλι θα μπορούσε κανείς να ε, κάνει συναλλαγές, άτυπες συναλλαγές, οι οποίες δεν μπορούν να ανοιχνευθούν σε σχέση με την, ε, προ... με την πρόταση να ε, διαγραφεί το υπερεθνικό σύστημα ε, αναγνώρισης συναλλαγών, νομίζω ότι αποτελεί ένα συμπλήρωμα της ΣΕΠΑ, αλλά αν υπάρξουν αλλαγές τότε θα αναδιαρθρωθεί ολόκληρο το σύστημα και δεν θα λάβουμε υπόψη δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα. Ως προς την εγκυρότητα αυτής της προσέγγισης θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ο κανονισμός θα πρέπει να συνεπάρξει με το επίσημο σύστημα ανείχνευσης συναλλαγών. Ε, δεν θα πρέπει να υπέλθουν αλλαγές ακόμα και αν θεωρούνται μικρές, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν, μάλλον να οδηγήσουν σε ε, λανθασμένη αντιμετώπιση του συστήματος ανείχνευσης ε, του συστήματος συναλλαγών. Επειδή ο κύριος Σίμων δεν είναι παρόν, ο κύριος που έχει το λόγο. Και εγώ θα σας δώσω το λόγο με τη σειρά μου, γιατί άκουσα τα σχόλια ε, θα τα λάβω υπόψη και θα συνεργαστώ με, με τον συνεισηγητή επί του θέματος, την συνεισηγήτρια και ελπίζω να φτάσουμε σε μία ε, εξισορροπημένη λύση και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επιτροπή για τα σχόλιά της. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου. Σας χαιρετώ και η Λίμπε θα συνεχίσει τις εργασίες της στις 2 το απόγευμα.